Απριλίου 1986. Είναι στη μνήμη μας πριν από 30 χρόνια κυρίες και κύριοι, στις 26 Απριλίου 1986 εξεράγει στην τότε Σοβιετική Ένωση, στην Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας, το μπλοκ 4 του πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ. Ε, υπήρξε πυρηνική σύνδεξη αυτό που αποκαλούμε μεγάλης έκτασης πυρηνικό ατύχημα που είχε τραγικές επιπτώσεις. Ραδινεργό υλικό εισήλθε στην ατμόσφαιρα. Μεγάλα τμήματα της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας μολύνθηκαν. Το ραδιενεργό νέφος πέρασε στην κεντρική Ευρώπη και μέχρι και τη Βόρεια Αφρική. Μέχρι σήμερα ο ακριβής αριθμός των ασθενών και ε, νεκρών λόγω των επιπτώσεων της ραδιενέργειας ε, δεν έχει καθοριστεί και είναι επίμαχος γιατί είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί. Αλλά κάποιοι υπολογισμοί για τις επιπτώσεις στην υγεία και για τους θανάτους ποικίλουν, αλλά όποια τάξη μεγέθους και αν ε, εξετάσουμε, οι τάξεις μεγέθους είναι δραματικές. Πολλές χιλιάδες λένε κάποιες εκτιμήσεις, ενώ άλλες ε, αναφέρονται σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Λιγότερο όμως θα ε, θυμόμαστε αυτούς ε, που χρειάστηκε να παρέμβουν για να αντιμετωπίσουν το ατύχημα. Ήταν νέοι άνδρες, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προστατευτικές στολές. Στάλθηκαν σε αυτό τον τόπο της καταστροφής για να την περιορίσουν. Σε αυτούς οφείλουμε το ότι δεν ήταν ακόμη πολύ χειρότερα τα αποτελέσματα του ατυχήματος. Πολλοί από αυτούς τους νέους, πολλοί από αυτούς τους ήρωες πλήρωσαν την ε, παρέμβασή τους με τη ζωή τους και την υγεία τους. Στην περιοχή χρειάστηκε να καταλήψουν ε, τις εστίες τους εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι, πολλές οικογένειες χρειάστηκε να επανεκατασταθούν, ολόκληρες κοινότητες καταστράφησαν και μέχρι σήμερα τα εδάφη και ε, τα τρόφιμα που παράγονται στην περιοχή είναι επιβαρημένα και πολλοί ακόμη υποφέρουν από τις συνέπειες. Ακόμη και τα παιδιά που γεννήθηκαν ε, πολλά χρόνια μετά από αυτή την καταστροφή. Το Τσερνόμπιλ παραμένει ως ερήπιο σίγουρα ένα μήνυμα, αλλά παραμένει και ένα πρόβλημα. είναι ιδιαίτερα δαπανερή η προσπάθεια να αποκατασταθούν τα κτίρια και η νέα ε, οικοδομή που θα πρέπει να την καταστήσει τον αρχικό τείχο προστασίας, ε, τον, αρχικό κλειό προστασίας που δημιουργήθηκε το 86 θα πρέπει να τελειώσει το 17 και θα κοστίσει 4 δις. Η αποφάση, οι αποφάσεις για την ε, χρήση πυρηνικής ενέργειας είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σίγουρα τα πυρηνικά νέφη και η ακτινοβολία δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα, γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα για την ασφάλεια και την πρόληψη. Και δεν πρέπει να περιοριστούν αυτέ τι προσπάθειε από εθνικά σύνορα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή η πυρηνική καταστροφή της, συγγνώμη, και η πυρηνική καταστροφή τη ε, Φουκουσίμα ε, η καταστροφή λοιπόν της Φουκουσίμα έγινε αίτιο για να υπάρξει έλεγχος της ασφάλειας 145 πυρηνικών εργαστασίων στην Ευρώπη. Πέρα από εθνικές ή πολιτικές διαμάχες, γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για την χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Αλλά πέρα από οποιασδήποτε διαφορές, πρέπει ούτως ή άλλως ακριβώς και λόγω της ε, μνήμης από αυτές τις καταστροφές πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη ε, πρέπει να είναι ασφαλή για το περιβάλλον τους. Αυτό είναι το αίτημα, αυτή είναι η έκκληση, αυτό είναι το καθήκον που πρέπει να εξαγάγουμε από αυτό το τρομερό ατύχημα του Τσερνόμπιλ πριν από 30 χρόνια και από την καταστροφή της Φουκουσίμα πριν από λίγα χρόνια. Αυτό το καθήκον, κυρίες και κύριοι, πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τη αντιμετωπίσει με την αναγκαία σοβαρότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την τιμή την δόκτωρα Αμάλ Αλκουμπάζη να συναντήσω, είχα την τιμή να τη συναντήσω είναι πρόεδρος του Κοινοβουλίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είναι προσκεκλημένη μας σήμερα και θέλω να την ευχαριστήσω, κυρία συνάδελφε.